Okay, well. Thank you Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε να ξεκινήσουμε. Σημείο πρώτο της σημερινής διάταξη έγκριση αυτής. Σας παρακαλώ φίλοι μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, η ημερήσια διάταξη ε, εγκρίνεται. Δεν βλέπω να υπάρχουν. Ανακοινώσεις του Προέδρου σημείο 2. Πρώτα απ' όλα έχουμε web streaming. Να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Και επίσης η εφαρμογή e-meeting είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη και τους βοηθούς των πολιτικών ομάδων από τις ταμπλέτες και τα λάπτοπ για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα έγκριση της ημερήσιας διάταξης, μάλλον έγκριση στο σημείο 3 των πρακτικών της συνεδρίασης της 11 η Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις στο τέλος, θα θεωρήσουμε εγκεκριμένα αυτά και να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία των εκθέσεων. Η κυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Πολύ σημαντική έκθεση των εισηγητών Τούρμες από τους Πρασίνους και της κυρίας Ριβαζή και πάλι από τους Πρασίνους. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω εδώ τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών Ήτρε και Έμβη, γιατί συνεργαστήκαμε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της Ενεργειακής Ένωσης και τη σύνταξη της έκθεσης. Να ευχαριστήσω και όλους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, ιδίω τον κύριο Μπούζεκ, τον πρόεδρο της Έμβη, και τους συνεισηγητές, τον κύριο Τούρμες και την κυρία Ριβαζή να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Όλαφ Χένκελ, αντιπρόεδρο, για να κάνει και εκείνος τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ο κύριος ε, Μπούζεκ είναι εδώ, <clears throat> μπορώ να πω εκ μέρους όλων, ότι του ευχόμαστε καλή επιστροφή και το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, ο φάκελος αυτός είναι πολύ σημαντικός με πολλούς σχετισμούς για τα ανανεώσιμα και για την οδηγία ενεργειακής απόδοσης που ψηφίσαμε στις 28 Νοεμβρίου στην Ήτρε. 1.700 τροπολογίες υπευλήθησαν στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι σημαντικότατη πρόκληση να αντιμετωπίσει κανείς ε, τόσο περίπλοκη πρόταση με τόσους πολλούς σχετισμούς με άλλες προτάσεις σε συνεδρίαση σε κοινή μάλλον συνεδρίαση επιτροπών. Να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή και όλους τους κοιόδης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άρα θα πάμε απευθείας στην ψηφοφορία. Οπότε, όσοι δεν έχουν καθίσει παρακαλώ να το κάνουν τώρα, 20 δεύτερα θα σας δώσω. In the meantime, push your cards in. <laughs> I hope we are all prepared. Για την ώρα κάντε μια δοκιμή. Ελπίζω να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, γιατί θα έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Πολύ ωραία, χωρίς έλεος, ξεκινάμε αμέσως. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 201. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πρώτη δοκιμή, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 24, 4 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Μάλιστα. Θα έχουμε εδώ πέρα αντιπαραθέσεις όπως βλέπω να ελέγξουμε. Well, Πέρας τις Ενεκρίθη. Σαράντα έξι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 501 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε, έστω να ελέγξουμε και αυτήν, όπως θέλετε. Πέρας, εγκρίνεται. Εντάξει τώρα, λέει ο πρόεδρος. Σαράντα εννέα, υπέρ. και αν εγκριθεί καταπίπτουν 502 και 503. Εγκρίνεται. «509 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «510 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία πενήντα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 512 υπέρ κατά να ελέγξουμε πέρας εγκρίνεται Περίπλοκοι συμβασμοί. Συμβαστική 3α ηλεκτρονικά. πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απεριφή. Συμβαστική 3B με ηλεκτρονικά. εγκρίνεται 5-16 υπέρ παρακαλώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 5-16 λέει πάλι ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε λοιπόν και εδώ Πέρας. Είχατε δίκιο. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. 50 και 5 και 7 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξετε. Ωραία. Ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Αυτή τη φορά είχα δίκιο τουλάχιστον. 518. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ζητήσετε έτσι κι αλλιώς έλεγχο, οπότε ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 5.19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Ε, ξανά. Υπέρ στην 5.19. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, εντάξει. Θα ελέγχουμε τα πάντα λοιπόν. Πέρας, εγκρίνεται. 5-20, υπέρ. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε λοιπόν. Πέρας, ίδια ακριβώς ε, πλειοψηφία. Ακριβώς ίδια. Το λέει και στα γερμανικά ο πρόεδρος. Συμβαστική 2α και θα πάμε απευθεία σε ηλεκτρονική ψήφο. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 11 σελίδα 12. Υπέρ. Σημαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα μου ζητηθεί να ελέγξω, οπότε ελέγχω. Πέρασε. Είχα δίκιο. Εγκρίνεται. Σελίδα 16 συμβαστική 4. Υπέρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5α ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας τώρα νομίζω, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. μπορούμε τώρα να υπερπηδήσουμε στη σελίδα 24 643 643 τροπολογία παρακαλώ υπέρ κατά τρο, ε, αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6α ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. Νέο άλμα στη συμβαστική 7 σελίδα 30. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 σελίδα 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 751 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε λοιπόν την 751 I close the vote. Yes, and it was rejected. Ωραία, απορρίφθηκε. 752 52 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε. 753 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε. Ωραία, α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. close. Πέρας. Rejected. 754 now. 754. 754. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Να είμαστε σίγουροι. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 755 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 756 υπέρ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 757 υπέρ κατά εποχές απορρίφθηκε. 758 υπέρ κατά εποχές απορρίφθηκε. 26 άγκρι υπέρ κατά εποχές ε, απορρίπτεται 759 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 760 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 761 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά is closed. Πέρας απορρίπτεται. 762 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 764 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 765 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 766 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται 767 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Όμως εντάξει ωραία ας το ελέγξουμε καλύτερα ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ Close. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. Πάμε στη σελίδα 39. 787. Τροπολογία 787. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 789. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. 9, let's check. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 789. Klaus. Πέρας. Απορρίπτεται. 790-791 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 792 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 793 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 794 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 795 υπέρ κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Α, καταπίπτει. Ναι, έχετε δίκιο. Uh, Πολύ ωραία. 5.13 και 7.96 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 803 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 805 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Closed. Adopted. Εγκρίνεται. 91. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εμένα μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Close. Adopted. Πέρας εγκρίνεται. Συνάδελφοι, ξέρω ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αλλά σηκώντε τα χέρια σας παρακαλώ. 811. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, εντάξει. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. And what is Closed. And it's rejected. Απορρίπτεται. 92 now. 4. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 812 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 8.13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8.15 υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη, καταπίπτει. 8.16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Close Πέρας. <laughs> And it is uh, rejected. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εντάξει, ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. And is closed. Πέρας. Adopted. Sorry. This... Εγκρίνεται. Συγγνώμη, αφήβρα είχατε δίκιο. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. All vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 8-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εντάξει, ωραία. Ας το ελέγξουμε. Close. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήσασταν τυχερός. Άγκρι 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 820 20 καταπίπτει, 8-21 υπερ κατά, αποχές, απορρίπτεται. και πάμε στην 8.32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές. Εμένα μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Close the votes. Ναι, είχα δίκιο. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στη σελίδα 50, συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται και πάμε στη σελίδα 52 συμβαστική 14 υπέρ σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά μου ζητάνε να ελέγξουμε οπότε ας ελέγξουμε δεν έχω αντίρρηση Πέρας. Και ατυχήσατε. εγκρίνετε. 8.85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Γιατί δεν βλέπω τα χέρια σας. Δεν τα σηκώνετε αρκετά. Τι να κάνουμε. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και ψηφίζουμε για την 885. Πέρας ψηφοφορία. Γι' αυτό πήγα σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Όχι, εντάξει, ας μην, ας μην ελέγξουμε και τη συμβαστική, ήταν σαφές. Συμβαστική 16, υπέρ, κατά, αποχές. Αυτήν όμως θα την, θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. And vote closed. Πέρας. Unfortunately it was adopted. Εγκρίνεται. 927, 928 together. 927, από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 929 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. Α, ναι, ωραία, ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Close. Πέρας. it was adopted. Ναι, εγκρίθηκε. 9.35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 και 9.30 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Πέρας εγκρίνεται. 9.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. What is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 9.34 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Closed. Πέρας της φοβορίας. Εγκρίνεται. 9.32, 9.33 καταπίπτουν και πάμε στην 9.36 και 9.37 από κοινού υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτονται. 9.43 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε. Close. Εγκρίνεται. Εκατόν είκοσι από κοινού υπέρ. Παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας όσοι είστε υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Α, απορρίφθηκε. Χάνουμε μια ομάδα τροπολογιών. Πάμε στη σελίδα 61. Περιμένω να γυρίσετε τις σελίδες και ψηφίζουμε την 9.74. Πάνσετ Γκερμπράντι Φέντρελι. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9.75 και 9.76. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9.77 υπέρ, κατά, αποχές Αγκρίνεται. 9.78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9.80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Αν και νόμιζα ότι εγκρίθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18α και 18b. Θα τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πρώτα τη 18α. Ηλεκτρονικός. 62. Σελίδα 62, 18α. Εντάξει, να σας περιμένω. 18α. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. 18α ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε και πάμε στη σελίδα 68 και ψηφίζουμε Τη βρήκατε. 1038. 1038 στη σελίδα 68. Σας περιμένω, σας περιμένω να το βρείτε. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να επαληθεύσουμε. Εψήφισαν άπαντες. Για βιαστείτε. Πέρας. Απορρίπτεται. 10.43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10.44. Υπέρ. Ε, τι να κάνουμε. Δεν θα την επαληθεύσουμε κι αυτή. Ήταν σαφέστατο. 10.44 υπέρ. 10.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Σελίδα 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά θέλετε οπωσδήποτε να ελέγξουμε, οπότε ας ψηφίσουμε και ηλεκτρονικός. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στη σελίδα 25. 23, συμβαστή 23, παρακαλώ είστε υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας, ευχαριστώ, υπέρ, κατά, αποχές, για να ελέγξουμε. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Α, απορρίφθηκε. 1106 υπέρ. Σελίδα 75. Πρέπει να πιάσουμε τις τροπολογίες της συμβαστικής. 1106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 11. Θέλετε παλήθευση. Πολύ ωραία λοιπόν να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 11.07. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζεται η υποψηφία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία για το πρώτο ήμιση και τώρα θα παραδώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο της Ήτρε. Ωραία. Να προχωρήσουμε. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να πάμε στη συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με διαφορά 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 28 άμεση με 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12.04. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Έλεγχο, έλεγχο. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 1207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1208 υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον πρέπει να επαληθεύσουμε. Δώδεκα άρχεται, πέρας, απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει λοιπόν να ελέγξουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφορία για την 39. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 12-10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 12-11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Όχι. 12-11. Άρχεται ψηφοφορία. Τι πάθατε. Θέλω να την κλείσω την ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 164 και 12-12 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-14 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Με συγχωρείτε, μόλις με διόρθωσαν, έπρεπε να έχω πάει στη 12-13, υπέρ, 12-13, υπέρ, κατά. Αποχές, νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε. 12-13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12-15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα 12-23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα να επαληθεύσω ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12-21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 12-22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12-24. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Επίσης απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. Εντάξει λοιπόν να επαληθεύσουμε 41 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 12.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα 12.49 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα. Unblock 167, 1256, 1257. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, μάλλον πρέπει να ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 1-6-8 και 1-2-6-1 ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12-65, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12-66, υπέρ, κατά, αποχές, και πάλι απορρίπτεται. 12-76, υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1268. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει. Να ελέγξουμε την 169. Άρχεται η Πέρας. Εγκρίνεται. 1271, 1272, 1273, 1274. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 1275. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφώς. Απορρίπτονται. Και τώρα συμβαστική 30. Υπέρ κατά αποχές νομίζω πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 31α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχιε του ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1406 μηδέν έξι. Πολλές σελίδες παρακάτω. Στη σελίδα μου είναι στην 82. Στην 102. 1406 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ο ηλεκτρονικός άρχεται την ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβεβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14.37 σας δίνω λίγο χρόνο, 14.35 στη δική μου σελίδα είναι στην 105, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14.39 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 14.40. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 14.41. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ξανά. 14.41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Για να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 1441. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1445. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να επαληθεύσουμε. 14.45. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Και τώρα από κοινού 184, 14.44, 44, 14, 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 14.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. Θέλετε έλεγχο. 14.43 η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 1446 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. 1446 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Καλά λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή, 186. 187, 187. Να συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 14-68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1482 και 1484 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 1483 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επαληθεύσω. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται 197. Πέρας. Εγκρίνεται. 1485 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία λοιπόν. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 1485 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41. Να ψηφίσουμε απευθείας ηλεκτρονικός, διότι φαίνεται ότι είναι επίμαχη. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 42 τώρα. Και πάλι θα ήθελα να ψηφίσουμε απευθείας ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1492 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία λοιπόν. 1492. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1494 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 43. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 14.95. Sorry. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1496 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 48 ηλεκτρονική ψηφοφορία. έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα 15-22 στη σελίδα μου 114. Σας δίνω λίγο χρόνο για να γυρίσετε τις σελίδες. 15-22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλά λοιπόν να ελέγξουμε 15-22 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 15-23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία λοιπόν, 15-23 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία και πέρας αυτής. Απορρίπτεται. Και τώρα συμβιβαστική 49 ηλεκτρονική ψηφοφορία, γιατί φαίνεται ότι θα υπάρξει μικρή διαφορά. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 50. Και πάλι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Συμβαστική 51. Και πάλι θα ήθελα να ψηφίσουμε απευθείας ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 1582. Στη σελίδα μου είναι 120 ε, η αρρύθμιση υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελεγξουμε 1522. άρχεται η ηλεκτρονική 1582. Πέρας εγκρίνεται. Και τώρα Πάμε στην 1586, λίγες σελίδες παρακάτω, σας δίνω χρόνο, Στη ε, ρύθμισή μου είναι 124 σελίδα. 1586. 1586 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά θα προτιμούσα να το ελέγξουμε, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, 16.24 και 16.25 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξω ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία 16.24 και 16.25. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 53. Ηλεκτρονικός ελεγχο παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία απευθεία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 16.33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16.34. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται μου φαίνεται. Καλά λοιπόν, να ελέγξουμε. 16.34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16.36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16.37 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 16.38 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 16.38. Πέρασε. Εγκρίνεται. 16.39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 1640 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξω τη 1640 πέρας εγκρίνεται 1645 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 1645 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 1647 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 1647 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 1646 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1648 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1649 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 1649 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 16.50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16.51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16.52 και 53 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Να ελέγξουμε λοιπόν 52 και 53 ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 16, 54 και 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξω λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για 54 και 55. Πέρας. Απορρίπτονται. 1657 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1656 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 1656. Πέρας εγκρίνεται 1659 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα Α, να ελέγξουμε λοιπόν 1659 το πρώτο τμήμα παρακαλώ πέρας απορρίπτεται Πολύ καλά που με βάλατε να το ελέγξω λοιπόν. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1660 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1661 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξω. 1661, 1661 η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 44, πάμε απευθείας ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 45 στην επόμενη σελίδα μάλλον, λέει ο Πρόεδρος, ή ηλεκτρονικά απευθείας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16.78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. 16.79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1680 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1681 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1682 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 46 ηλεκτρονικά, πέρας, Εγκρίνεται. 16, 86 και 87 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 16, 88 και 89. Και 16, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 16, 91 και 1662 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 1693 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε λοιπόν τη 1693 παρακαλώ. Πέρα. Ζητώ συγγνώμη και διορθώνω. Εγκρίνεται 1694 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 47. Απευθείας ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 1699 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17.00. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε συμβαστική 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 2.18 και άγκρι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε τη 2.19 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 55 εγκρίνεται. 2, 7 αιτιολογική υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2, 28 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2,40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.62 υπέρ. Κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε τη 262 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτε. Συμβαστική 59 υπέρ. Μάλλον ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική 8 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξω την 8 για την αιτιολογική 6. Εγκρίνεται. Και πάμε στην επόμενη σελίδα 268 στο κείμενό μου απορρίπτεται 269 στο συγγνώμη λέει ο πρόεδρος η 268 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρασε εγκρίνεται 269 υπέρ δεν βλέπω χέρια κατά τώρα βλέπω χέρια απορρίπτεται λοιπόν 2.71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.74 υπέρ. Κατά. Είπε πρώτα απορρίπτεται και μετά αποχές. Ο πρόεδρος διόρθωσε απορρίπτεται. Συμβαστική 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 61 απευθείας ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 2,77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λέει ο Πρόεδρος. Ναι, άγκρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. Συμβαστική 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 289 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 66 υπέρ. Όχι ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. οκτώ υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 308. Παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 339 αιτιολογική 17 μαζί με άγκρι 8 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτε. 341 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 341 παρακαλώ. Πέρας. εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.48 υπέρ. Παρά, ε, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβαστική 72 απευθείας ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρασε. εγκρίνεται. Συμβαστική 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε. Στην 369. Σαλίδα 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 74. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην συμβαστική 75 στην σελίδα 148. Συμβαστική 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 389 αιτιολογική 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφορία από τις 26 πέρας is accepted. εγκρίνεται και πάμε στη τελική σκέψη 23 390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 76 λέω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ Πέρας. Απορρίπτεται. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 393 και άγκρι 10 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 394 όχι συγγνώμη, 395 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 396 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε στη συμβαστική 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην... Στην τροπολογία 404 στην 150 στο δικό μου έγγραφο. Περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αν ελέγξουμε, εντάξει, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία 404. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση οφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 79, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε, άγκρι 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 82, να, το, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά απευθείας, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, για την τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 82 εγκρίνεται. Συμβαστική 83 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 84 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 85 να ψηφίσουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τώρα, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 86 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 87. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά απευθεία. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Όχι, τώρα. Ολοκληρώθηκε. εγκρίνεται. 4.39 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 4.40 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 88 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 89 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 447 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 448 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 448 τώρα. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 91 υπέρ, κατά, απο... αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 456 υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ε, τροπολογία 456. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 455 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 461 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 93 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 465 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να το ελέγξουμε, να είμαστε βέβαιοι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 465. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίπτεται. Λοιπόν, και τώρα ψηφοφορία unblock από το 202 στο 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται όλες αυτές και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση ψηφίστε παρακαλώ τώρα ηλεκτρονικά The vote is closed. περασε ψηφοφορίας 61, So <laughs> What? congratulations. Maybe the rapporteurs want to say few words. Yeah. Well, first of all, big... calm down, ladies and gentlemen. Καταρχάς, ας ηρεμήσουμε. Ψυχραιμία. Να συγχαρούμε τους συνεισηγητές. Θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι. Θα ήθελα εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω τους αντιπροέδρους της Ήτρε, εσάς αγαπητέ συνάδελφε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Ιανουάριο του 2018 και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία.